Ladies, gentlemen, colleagues, shall we get started? Ξεκινάμε αγαπητοί συνάδελφοι. The agenda, you have draft agenda. Έχετε ενώπιόν σας την ημερησία διάταξη. Έχουμε ένα πρόβλημα με το θέμα γενικευμένων προτιμήσεων και είχαμε πει να, απο... να αναβάλουμε την ψηφοφορία και και το θέμα αυτό μάλλον θα έρθει στη μέση διάταξη μόνο στις 3 Μαρτίου. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν να γίνει αυτή η αλλαγή, να το βγάλουμε από τη μέση διάταξη, θα αποφασίσουμε όμως αργότερο. Υπάρχουν, ε, πέραν αυτού υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις, προτάσεις τροποποίησης στη μέση διάταξη. ως συνήθως. Έχουμε ένα ναι. κατάλογο της αλληλογραφίας που έχουμε λάβει και αν σας ενδιαφέρει κάποιο θέμα μπορείτε να ζητήσετε να τα δείτε από τη γραμματεία. Περνάμε στο σημείο 3, το πρώτο ουσιαστικό θέμα. περαιτέρω χρηματοδοτική μακροοικονομική συνδρομή στη Γεωργία. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ο υποφαινόμενος συνεισηγητής και η άποψή μου είναι εξής. Η Κομισιόν προτείνει περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Γεωργία να χορηγηθεί. 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οΐμιση αυτού του ποσού <clears throat> σε χορηγήσεις και το άλλο μισό σε δάνεια. Όπως θυμόσαστε, οι τελευταίες προτάσεις αυτού του είδους είχαν παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής μας για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. και θέλαμε η Κομισιόν να μας ε, παρουσιάσει τα πορίσματά της σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της βοήθειας και την διαφάνεια και λογοδοσία αυτής της ε, βοήθειας. Και η Κομισιόν αυτή τη φορά ακολούθησε αυτό που είχε αποφασίσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά και το κείμενο τη πρόταση τη Κομισιόν για χρήματα οικονομική συνδρομή στην Γεωργία. ευθυγραμμίζεται απόλυτα η πρότασή της με τις προηγούμενες αποφάσεις μας στην περίπτωση της Ουκρανίας αλλά και της Μολδαβίας. Για τους λόγους αυτούς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να εγκριθεί βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας. Μη όντως λόγου για να ακολουθήσουμε τις ε, άλλες διαδικασίες πέραν της Ουκρανικής και Μολδαβικής. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση της Κομισιόν. Αυτό είναι η πρότασή μου λοιπόν σε εσά να εξετάσουμε το κατά πόσο θέλουμε να ακολουθήσουμε την απλοποιημένη διαδικασία άνευ τροπολογιών. Για να μην χρονοτριβούμε λοιπόν, Γνωρίζω ότι η μέση διάταξή μας είναι πεφορτωμένη. Και σας δίνω το λόγο για να μου δώσετε μια απάντηση στην πρόταση να προχωρήσουμε με την απροποιημένη διαδικασία. Ο κύριος, κύριος Γκέρνς. Παρά την πρότασή σας για την απλοποιημένη διαδικασία, έχω να κάνω δύο απλά σχόλια για το περιεχόμενο και για τη διαδικασία αντιστοίχως. Δεδομένου του ότι η κυβέρνηση της Γεωργίας θεωρείται πλέον συνυπεύθυνη για τον πόλεμο του 2008 με τη Ρωσία, μήπως μπορούμε να έχουμε την εξασφάλιση ότι δεν θα πάνε τα χρήματα αυτά, ούτε κάποιο τμήμα τους, για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δαπάνες της Γεωργίας. Μήπως μπορούμε να έχουμε αυτή την διαβεβαίωση από την Κομισιόν. Και θα μπορούσε η Κομισιόν να μας πει ποια είναι η κατάσταση της απορρόφησης και της εκταμείευσης του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια για αυτό το κονδύλιο. Επίσης, το Κοινοβούλιο στην ε, αιτιολογική του έκθεση για τα θέματα αυτά 2008 ζήτησε πιο τακτικέ εκθέσει από την Κομισιόν σε εμά για τι χρηματοδοτικές αυτέ ενέργειε. Αναρωτιέμαι αν αυτό έγινε πραγματικότητα. Τέλο, διαδικαστικά <clears throat> για τα θέματα διαδικασία. Σαν νέο μέλος αυτής τη Επιτροπής βλέπω λιγάκι παράλογο το να αντιμετωπίζουμε κάθε συμφωνία χρηματοδοτικής αρρωγής ως ένα έκτακτο μέτρο το οποίο πρέπει να περάσει μια διαδικασία ad hoc. Ενώ είναι τόσο συνηθισμένε αυτές οι αιτήσει για χρηματοδοτική αρρωγή, μήπως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να δημιουργήσει και μία συμφωνία πλαίσιο, ένα πλαίσιο συμφωνίας, ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά ξεκινάμε από το μηδέν για κάθε μία από τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Άλλες παρατηρήσεις πρωτού ζητήσω την άποψη της Κομισιόν. Όχι η Κομισιόν. Ο κύριος Πρόεδρος, Τεμπράνο. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την ερώτησή σας, θα ήθελα να σας καθησυχάσω και να σας πω ότι τα χρήματα του NFA χρησιμοποιούνται για έρευνα και ε, για εξισορρόπηση της οικονομικής χρήσης. Δεν θα δοθούν σε καμία περίπτωση για ενίσχυση του προπολογισμού. Υπάρχει πολύ σημαντική ε, διαδικασία διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τώρα τα έκτακτα αυτά μέτρα, ναι, είναι έκτακτα τα μέτρα. Αυτή τη μορφή η συνδρομή είναι έκτακτη μορφή. Έχουν παρουσιαστεί κάποια πράγματα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάρα πολύ ε, σοβαρά στην ε, παρουσίαση μιας πρότασης ε, ε, κανονισμού πλαίσιου που θα παρουσιαστεί ε, πολύ σύντομα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Βάσει του χρονοδιαγράμματός μας η παρουσίαση θα γίνει το Μάρτιο μάλλον. Υπήρχε και η ερώτηση για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα υπόλοιπα NFS. Συγγνώμη, δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα την ερώτηση αυτή. Η ερώτηση ήταν... Αν για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ε, μικροοικονομικής ε, συνδρομής ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξελίξεις. Φυσικά κύριε Πρόεδρε, απαντά η Επιτροπή, ω συνήθω θα παρουσιάζουμε μια ετήσια έκθεση για την εφαρμογή τη μικροοικονομική συνδρομή. Ε, αυτό θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο πριν από τον Ιούνιο. Όσον αφορά τώρα τη Μολδαβία, ε, να ανακοινώσω ότι έχει δοθεί η πρώτη δόση και για την Ουκρανία Ακόμα συζητάμε τους όρους αυτής της διαδικασίας. Ε, δεν ήταν εύκολη συζήτηση. Έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος τις τελευταίες εβδομάδες. Ακόμα εκρεμεί ένα θέμα το οποίο θεωρείται σημαντικό από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα σα ενημερώσουμε στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή τη μικροοικονομική ε, συνδρομή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Φαίνεται ότι Πλέον έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την πρότασή μου, θεωρούμε ότι εγκρίνεται χωρίς ενστάσεις. Χωρίς καμία τροποποίηση. Moving to item Να περάσουμε τώρα στο σημείο 4. Ένωση καινοτομία. Mm. Μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση. Mm. Όπως γνωρίζουμε, μία από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική του 2020 είναι η Ένωση Καινοτομίας υπεύθυνη για την έκθεση επί είναι η Ήτρε και η Επιτροπή μας αποφάσισε να παρουσιάσει και μία γνωμοδότηση. Η συντάκτρια είναι η Νέζε Βάιντερη από το ΕΛΚ. Δεν είναι παρούσα σήμερα. Ο κύριος Κάσπαρη θα την αντικαταστήσει. Έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, δεν την αντικαθιστώ. Θα διαβάσω όμως ε, τα όσα μου έδωσε. Η κυρία Βαϊντερέ μου ζήτησε να διαβάσω το εξής. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία μου κατά τη δεύτερη αυτή ανταλλαγή απόψεων για τη γνωμοδότηση. Είχα ανηλμένε υποχρεώσεις ε, για την ε, δεύτερη συνεδρίαση καινοτομίας και συνεργασίας στο Ισραήλ για την Ένωση Κοινοτομίας αποφάσισα να σταθώ και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στην έκθεση της Επιτροπής ΣΥΤΡΑ η οποία θα εκφράζει την τελική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λυπάμαι που δεν έχουμε λάβει ακόμα το σχέδιο κειμένου ε, ούτε και κάποια προστίκη στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ΣΥΤΡΑ ε, και το μόνο που έχουμε είναι κάποια στοιχεία που λάβαμε πριν από την πρώτη μας ανταλλαγή απόψε τον Ιανουάριο. Θα ήθελα να σταθώ και στα δύο αυτά κείμενα. Η Ήτρε μου είπε ότι θα μου δώσει το πλήρε σχέδιο έκθεση του αύριο και γι' αυτό ακριβώ έχουμε και μία έκτακτη παράταση για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι την Παρασκευή για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και τα δύο κείμενα. Δεδομένων των συνθήκων θα παρουσιάσω και εγώ αρκετέ τροπολογίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να ανταγωνίζεται με χώρε όπω είναι η Κίνα για τι τιμέ παραγωγή το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα έγκυται στην κοινοτομία, στις τεχνολογικές μας δυνατότητες και στις ε, δυνατότητες που έχουμε εν γέννη. Θα υπάρχουν άμεσες και έμεσες επιπτώσεις ε, για το διεθνές εμπόριο και είναι σαφές ότι η σαφής επίπτωση της κοινοτομίας ε, μπορεί να γίνει μέσω αύξηση τη Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα ανά τον κόσμο, κυρίως ενώπιον τη κίνα ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ιαπωνία, διότι έχουν ανταγωνιστικέ τιμέ, ευνοϊκή νομοθεσία και ε, προηγμένη τεχνολογία. Από το έγγραφο που σας έχω διανέμει θα δείτε ότι έχουμε ελάχιστη προστασία της Ευρωπαϊκής Πνευματικής Οδιοθεσίας ε, ιδιοκτησίας της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας και τη μεταφορά τεχνολογίας σε τρίτες χώρες. Οι τιμέ θα πρέπει να μειωθούν για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να μπορέσουμε να έχουμε και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για του Ευρωπαίου ερευνητέ. Από πλευρά εμπορίου και μόνον, η καινοτομία θα πρέπει να έγκυται σε εταιρικέ σχέσει εμπορίου που θα ε, βασίζονται στην αμοιβαιότητα και στον θεμητό ανταγωνισμό. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι οι ευνοϊκέ συνθήκε εμπορίου ε, και οι τιμέ θα πρέπει να ισχύουν ε, και για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς και για να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας θα πρέπει να το θέσουμε αυτό ως προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε πολιτική και οικονομική στήριξη και η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασίζεται στην πράσινη οικονομία και σε άλλους τομείς και δεν θα πρέπει να χάνουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα δίνουμε και τη χρηματοοικονομική στήριξη για να έχουμε καινοτομία σε διάφορου τομεί και θα υποστηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσει, διότι είναι η βασική οικονομική παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήθελα να διαβάσω κυρία Βάιτερε. ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι διαβάσατε τα σχετικά στους φακέλους σας. Μήπως υπάρχει κανένα σχόλιο ο Βίλιαμ Μπάρτμοθ. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι πρόλαβα να το διαβάσω σε βάθος, αλλά ήθελα να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Θα μπορούσα να κάνω και 22, αλλά θα κάνω μόνο δύο. Για να μπορέσει η Κομισιόν να απαντήσει με συνέπεια επί των κυρίων θεμάτων. Λοιπόν, τα εξής. Ένα γενικό, ένα ειδικό. Πρώτα το γενικό, μετά το ειδικό. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσει κανείς για την καινοτομία. Δεν γίνεται, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτό αντιτίθεται και αντιστρατεύεται την εμπειρία που είχαμε με την καινοτομία τα τελευταία 100 χρόνια. Η Κομισιόν πιστεύει ότι μπορεί. Τι είναι ρωτό λοιπόν. Πώς θα νομοθετήσει για καινοτομία. Γιατί νομίζετε ότι μπορείτε. Και το δεύτερο θέμα τώρα που είναι πολύ λιγότερο γενικό. Πριν να εκλεγώ είχατε καταθέσει την προσωρινή οδηγία για τους εργαζόμενους που κατέστησε πιο δύσκολο πιο δύσκολη την προσωρινή εργασία και πολύ πιο δύσκολο για τους εργοδότες να απασχολήσουν μερικώς άτομα. Ενώ αν θέλουμε καινοτομία πρέπει να έχουμε μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση οποιοδήποτε θέλει να καινοτομήσει θα χρειαστεί να δουλέψει μερικός για κάποιον άλλον για να έχει το χρόνο και για να κάνει τα ψώνια του κλπ. Έτσι μόνο θα μπορέσει να καινοτομήσει στον ελεύθερο του χρόνο. Και πολλές από αυτές τις καινοτομίες μπορεί να μην λειτουργήσουν τελικά, αλλά άλλες μπορεί να είναι το καινούριο Google, η νέα Microsoft, σαν microsystems και άλλα τέτοια πράγματα. Τα μικροσυστήματα του ηλίου δηλαδή. Ελπίζω να απαντήσει η Κομισιόν ε, ρητά, όχι όπως πάντα να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Να το σκεφτεί και να μας δώσει μία απλή απάντηση. Γιατί θέλει να καταστρέψει την καινοτομία νομοθετώντας πάση θυσία. Συστηματικά μάλιστα και την οδηγία της προσωρινής εργασίας και την καινοτομία δεν τα καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω στον αγαπητό μου συνάδελφο. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά κάποια δισεκατομμύρια ευρώ σε θέματα έρευνα και καινοτομία, το ερώτημα είναι τι θέλουμε να υποστηρίξουμε και προ θα πού να κατευθύνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία μετά την κρίση. Σε όλη την οικονομική ιστορία από την εποχή των ασυροχαλδαίων υπήρχαν πάντα παρεμβάσεις από το κράτος, από το κοινωνικό σύνολο αν θέλετε, για να υπάρξει ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών ή κοινωνικών τομέων. Για μένα, για την περίοδο μετά την κρίση, είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε μέχρι τώρα. Και να μπορέσει να εξασφαλίσει να έχει μια οικονομία η οποία εν μέρει είχε να πόδι στο παρελθόν και εν μέρει είχε να πόδι στο μέλλον. Αναφέρθηκε παραδείγματο το παράδειγμα τη πράσινη οικονομία. Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι κάνουν οι κύριοι οικονομικοί μα εταίροι, τι κάνουν οι Κινέζοι, τι κάνει η Νότια Κορέα, τι κάνουν τα κράτη στην ε, Αμερικανική Ήπειρο για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Σίγουρα τους ενδιαφέρουν οι ανανεώσιμες ενέργειες, οι εξοικονομίες ενέργειας, οι πράσινες οικονομίες. Όλοι αυτοί είναι οι τομεί όπου θεωρούμε ότι εκεί θα υπάρξει η πηγή της ανταγωνιστικότητας για αύριο. Πρέπει λοιπόν να κατευθύνουμε την οικονομία μας προς τέτοιου είδους τεχνολογίες, προς τέτοιους οικονομικούς κλάδους και βέβαια από τη στιγμή που μιλάμε για πράσινες τεχνολογίες μιλάμε για καινοτομία <clears throat> και πρέπει να θέσουμε το ερώτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας και του καθεστώτος προστασίας της καινοτομίας. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ αυστηρό καθεστώς για τις ε, ευρεστεχνίες ή ένα σύστημα το οποίο δίδει το, τη σωστή ανταμοιβή στην καινοτομία αλλά επιτρέπει στο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Παραδείγματος χάρη για τις τεχνολογίες αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ, Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να μιλήσω εξ ονόματος ε, του σκιώδης εισηγητού μας από τη δική μας ε, ομάδα, του Τζο Higgins, ο οποίος είναι μέσα στα, είναι ως τα αυτιά στη διαδικασία εξόδου από την κρίση μέσα στην προεκλογική εκστρατεία στην Ιρλανδία. Και μου είπε σημεία τα οποία θα ήθελε να αναφέρω και θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε την αλληλοσύνδεση μεταξύ οικολογικών και κοινωνικών θεμάτων. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει <clears throat> ότι για να βγούμε από την οικονομική κρίση, μάλλον όταν έρθει το τέλος της οικονομικής κρίσης, το οποίο δεν το βλέπουμε ακόμα, οι πολιτικές καινοτομίε θα πρέπει να συμβάλλουν στο να ξεπεράσουμε την ανεργία, τα προβλήματα τα οποία έχουμε στον κοινωνικό τομέα κτλ. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν με ποιο τρόπο αυτές οι πολιτικές θα συμβάλλουν για την υπερπίδηση αυτών των εμποδίων που αποκλείουν όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών από τον παραγωγικό ιστό των χωρών μας. Και διάβασα σήμερα μια επιστολή από τον Γερμανό γραμματέα του Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργατικών ενώσεων προς την Επιτροπή ΑΦΚΟ όπου είπε ότι ο φορέας του δεν θα υποστηρίξει μια πλήρη αλλαγή των συνδικών σε σχέση με τον μακροχρηματοοικονομικό έλεγχο και ούτως θέλω να συνδέσω τη συζήτηση που έχουμε στις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εστιαστεί η προσοχή όλων και της Κομισιόν και των κρατών μελών όμως, ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια κατεύθυνση της καινοτομία ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ο Τζο Higgins θα σας δώσει εν καιρό κάποιες τροπολογίες συγκεκριμένες που θα καταθέσει σε αυτή την έκθεση και φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε στη συνέχεια να τη συζητήσουμε στην περαιτέρω εξέταση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα λάβει το λόγο. Γεια σας. Θα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι ο επικεφαλής ε, του τμήματος από την αρμόδια υπηρεσία δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα και θα σας απαντήσει γραπτός. Έχουμε σημειώσει τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να υπάρχει λόγος για την απουσία του. Το γεγονός ότι δεν είναι κανείς ε, εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει για το θέμα αυτό, ελπίζω να δικαιολογείται, γιατί αυτό είναι ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει και σχέδιο έκθεσης, γνωρίζετε και το χρονοδιάγραμμά μας. Απαράδεκτο το θεωρώ να μην μπορεί να έρθει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει. διότι ήταν αναμενόμενο να υπάρχουν ερωτήσεις στις οποίες θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί προηγούμενο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε απαντήσεις γραπτός στις επόμενες ημέρες ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα διαδικαστικό θέμα, επιτρέψτε μου Πρόεδρε, με την ε, συνήθεια ευλωτία σας μου πήρατε τα λόγια από το στόμα αυτό το οποίο θέλατε να πείτε είναι ότι εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπή του Κοινοβουλίου που ελέγχει αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το γεγονός ότι δεν έρχεται κανείς χωρίς να μας εξηγείτε γιατί ε, είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν είναι εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν συγκεκριμένες φυλές που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα έπρεπε να θεωρούν ότι ε, τους υποτιμάτων να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Όλοι έχουμε ερωτήσεις, ε, αλλά το θέμα είναι... Αλλά ούτε καν ε, λέμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τι έχει πια στο πρόγραμμά του ο οποιοδήποτε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορεί να έρθει εδώ να απαντήσει στην Επιτροπή μα και δεν μπορεί να παραστεί. Ίσως θα μπορούσα να διαβιβάσω λοιπόν και το ερώτημα μέσω του Προέδρου. Γιατί δεν μπορεί να έρθει ο λόγο κύριος. Πρόεδρος. Ίσως να είχε κάποιο ατύχημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην μπόρεσε να είναι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, έστω ότι δεν παρέστη ο εκπρόσωπος λόγω ενός πολύ πολύ σοβαρού ατυχήματος. Ίσως θα έπρεπε να του διαβιβάσουμε λοιπόν αυτού του απόντος ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για το ατύχημά του και να το ευχηθούμε καλή ανάρρωση το συντομότερο δυνατόν για οποιοδήποτε ατύχημα είχε. Ο κύριος Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφέ ότι δεν πληροφορηθήκατε ούτε εσεί ούτε η Γραμματεία για το γεγονό ότι η Κομισιόν θα ερχόταν, ότι δεν θα ερχόταν γι' αυτό το σημείο τη ημερησία διάταξη. Μπορεί να είναι ένα ατύχημα, μπορεί να είναι μια καθυστέρηση. Εγώ προτείνω να αναβάλουμε την εξέταση αυτού του σημείου, να το θέσουμε στην τελευταία σειρά στην ημερησία διάταξη. Μήπω η Κομισιόν χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία να στείλει κάποιον ο οποίο μπορεί να απαντήσει για το θέμα αυτό. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση. Απλώς να διευκρινίσω το εξής. Ε, ο κύριος Δεγκράφ, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τα θέματα πολιτικής καινοτομίας, δεν μπόρεσε να παραστεί και εγώ είμαι υπεύθυνη για να καταγράψω τις ερωτήσεις του και θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείται σε ευθέτω χρόνο, λέει ο πρόεδρος ε, υποθέτω ότι χρόνος ήταν σήμερα, η σημερινή μέρα. Okay. We take... Καλά, καλά. Καταγράφουμε αυτήν την ε, κατάσταση πραγμάτων. Τι είναι αδυναμία της Κομισιόν να είναι παρούσα για το θέμα αυτό. Ε, κάποια σχόλια από τον αντικαθιστώντα την εισηγητή, την εισηγήτρια. Προθεσμία τροπολογιών στις 14 του μηνός, στις 6 το απόγευμα. Ας πάμε στο σημείο 5 όμως. Εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και η ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Απασχόλησης που είναι η επί αρμόδια επιτροπή. Όπως ξέρετε, πέρσι εμεί εγκρίναμε μια έκθεση πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μας για ένα παρόμοιο θέμα. Εύλογον θα το επομένως να συμβάλλουμε και στη διαμόρφωση της έκθεσης αυτής της Επιτροπής Απασχόλησης επειδή είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος αυτό το θέμα, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης που είναι στο φάκελό σας. Η κυρία Τοκία Σαΐφη είναι η συγγήτρια και Τοκία έχει το λόγο. σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για τη φωνή μου που είναι λίγο σπασμένη αλλά είμαι κρυωμένη. Ήθελα να έρθω σήμερα το απόγευμα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που φέρω την ευθύνη αυτή τη γνωμοδότηση, κάτι που μου επιτρέπει να συνεχίσω τι εργασίε τη Επιτροπή μα, για συνεχίζοντα από την έκθεσή μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου και τα κοινωνικά δικαιώματα στι διεθνεί συμφωνίε. Θέλω να ακολουθήσω την ίδια συνενετική μέθοδο όπω και στην έκθεσή μου, γι' αυτό το κείμενο που σα υποβάλλω είναι πάρα πολύ σύντομο κάποιες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη του να ενισχύσουμε το ρόλο των αρμοδίων διεθνών οργανισμών και επίσης την συνεργασία μεταξύ αυτών των διεθνών φορέων. Παραγματος χάρη, ο ΠΟΕ και το, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας θα πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσουν να έχουν την απόλυτη υποπτία των εργασιακών θεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ΔΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΣΑ UNESCO. Είναι μια σειρά φορέων που μπορούν να επιληφθούν του θέματος αυτό. Θεωρώ επίσης ότι είναι απαραίτητο να τεθεί και μια ρήτρα εταιρική ευθύνη σε όλες τις συμφωνίες που ε, διαπραγματεύεται η Κομισιόν και η έκθεση του κ. Χαλέμ Ντεζίρ τον προηγούμενο Νοέμβριο δείχνει ότι αυτή η άποψη έχει ευρεία υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι και τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν κατανοήσει το γεγονός ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πάντα αυτή η ρήτρα για την εταιρική ευθύνη. Θέλω να αναφέρω επίση την περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι γεγονό ότι οι μεγάλε ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ έχουν να δώσουν μια σημαντική συμβολή στην μεταλαμπάδευση των ευρωπαϊκών αρχών και τη κοινωνική ευθύνη των εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά οποιαδήποτε εταιρεία, μικρή, μεγάλη ή μεσαία, θα έχει και αυτή η μεγάλη ευθύνη για να το επιτύχει αυτό. Βέβαια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνει πολύμορφες εταιρείε με διαφορετικές δραστηριότητε, αλλά το θέμα της προώθηση της κοινωνική ευθύνης είναι πολύ σημαντικό για όλες αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Εγώ προσπάθησα πρώτα απ' όλα να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν η οποία προετοιμάζει μια ανακοίνωση για την παγκοσμιοποίηση της δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δεν πρέπει η Κομισιόν να αγνοήσει το θέμα αυτό. Μένουν δύο θέματα ακόμα εκκρεμή. Καταρχήν το θέμα του εθελοντικού χαρακτήρα ή αντίθετα δεσμευτικού για την κοινωνική εταιρική ε, ευθύνη. Το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής έχει πάντα στραφεί κατά της ε, υποχρεωτικότητος της ε, ρήτρας αυτής, της χρησιμοποίησης αυτής της ρήτρας Μήπω τώρα πρέπει να αλλάξουμε άποψη και ίσω πρέπει να διευρύνουμε αυτή την κοινωνική ευθύνη και στα θέματα που είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Τι γίνεται με τι διμερείς συμφωνίε και τι γίνεται αν αυτή η ρήτρα δεν τύχει σεβασμού από κάποιον από του εταίρου μα. Και αυτό τίθεται φυσικά το ερώτημα και στα πλαίσια του γενικευμένου συστήματο προτιμήσεων. Ποιε είναι οι κυρώσει σε περίπτωση παραβίαση αυτή τη ρήτρα μέχρι στιγμή έχουν σταθεί ιδιαίτερα περιορισμένε. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε και κλείνουμε αυτό το τόσο σημαντικό σημείο η Κομισιόν να παρακολουθήσει αποτελεσματικά την εφαρμογή της ρήτρας αυτής και να ξέρουμε τι θα γίνει σε περίπτωση μη σεβασμού της. Ήταν πάρα πολύ σαφή αυτά που είπατε. Το ΚΙΑ. είναι το λόγο σε όσους θέλουν να λάβουν το λόγο. Ε, ε, ε. Ε, μου είπαν ότι σκιώδης συγητής του ΕΡΚ είναι στην Αφρική. Ο κύριος Σόλτς από την Κούγα έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα πάω στην Αφρική, στον Τακά, στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονό ότι κάνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Α, η εισηγήτρια είναι η, η, δίκη, η από την άλλη ομάδα, είναι ήδη. Χαιρετίζω ιδιαίτερα λοιπόν αυτή την ευκαιρία συζήτηση. γιατί αντιμετωπίζει μια σημαντική αίτηση αυτή η έκθεση που πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω την συντάκτρια γνωμοδότησης για την παρουσίαση της γνωμοδότησής της αλλά η ομάδα μας έχει κάποιες παρατηρήσεις και ενδεχομένως θα καταθέσουμε και τροπολογίες οι οποίες με έναν τρόπο κριτικό <clears throat> και εκπεφρασμένο θα θέλουν να τονίσουν ότι στο παρελθόν δεν ήταν επαρκής η αυτορύθμιση στα θέματα αυτά, δηλαδή η εθελοντική κοινωνική εταιρική ευθύνη. Θυμάστε ίσως τα προβλήματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν με την παραγωγή σοκολάτας από την ακτή ελεφαντοστού που ενέπλεξε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείε σε συνθήκες οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Η κατάσταση λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων και των υπεργολαβικών τους εταιρείε δείχνει <clears throat> ότι αυτό το θέμα αφορά ε, όλο τον κόσμο και σε σχέση με αυτό οι ευρωπαϊκές εταιρείες στο παρελθόν δεν έχουν πάντα κρατήσει μια σωστή στάση. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει σαφείς κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ρήτρες αυτού του είδους. Και προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν θα κινηθούμε ως πολιτική ομάδα και πιστεύω ότι και στις περαιτέρω συζητήσεις για αυτή την έκθεση θα πρέπει να τονιστεί εκπεφρασμένα η ευθύνη των ε, επιχειρήσεων, η εταιρική ευθύνη και θα πρέπει να τονιστεί η ανάγκη αυτή η εταιρική ευθύνη να ελέγχεται αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε αυτές εργάζονται για τη βελτίωση του εργασιακού και βιωτικού καθεστώτος στις χώρες όπου εργάζονται. Ευχαριστώ. Yes. <laughs> Double name. <laughs> Eh, e <laughs> Διπλό όνομα έχω. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πριν γίνω ευρωβουλευτής, εγώ ήμουν στις δημάσιες υποθέσει για τι ε, μεγάλε οικονομικές ε, επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να υιοθετήσουν πολιτικές εταιρική κοινωνικής ευθύνης για να αυτοπροβληθούν, να πούν κάποια πράγματα για τη μάρκα τους, για τον κώδικα διοντολογία τους, για τις αξίες τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους το επιβάλλουμε, διότι έχει αξία μόνο όταν υιοθετείται κατά συγκεκριμένο τρόπο από αυτές τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να περιμένει επί εθελούσιας βάσεως οτιδήποτε άλλο δεν είναι χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη φορά έχουμε εκπρόσωπο, τη Μαγδελένα Ρούντα. Παρακαλώ. Κριστίν Τράιμπερ. <laughs> Επικεφαλή του Τμήματο Απασχόληση και Διεθνών Υποθέσεων. Χαιρόμαστε που ασχολείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το θέμα αυτό τη κοινωνική διάσταση τη εταιρική κοινωνική ευθύνη και το γεγονό ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είμαστε υπέρ του διαλόγου στον τομέα τη απασχόληση και των κοινωνικών υποθέσεων και ε, σε διμερές επίπεδο με του εταίρου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώ. Όπως ακούσαμε, είμαστε υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τους στόχους απασχόλησης, ε, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνάδουν και με τους κοινωνικούς στόχους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, και τις ε, κυβερνήσεις. Θα συνεχίσουμε να είμαστε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοπρεπούς εργασίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω εμπορικής πολιτικής και κυρίως των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ε, να κυρώσουμε και να τηρούμε τη σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας καθώς και άλλες συμβάσεις που μπορεί να επικαιροποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Όσον αφορά τώρα τις συμφωνίες εμπορίου, το θέμα συζητήθηκε στα πλαίσια του ψηφίσματο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι διεθνεί προδιαγραφές για τι εμπορικέ συμφωνίε. Δεν θα ήθελα να επανέλθω διεξοδικά επί του θέματος αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εμένει στη θέση της ότι ένα σύστημα που βασίζεται στο διάλογο με τις χώρες εταίρους και το γεγονός ότι θα πρέπει να δεσμεύονται με τις υποθέσεις αυτές είναι πολύ καλύτερο από το να τους αναστέλλονται κάποια συγκεκριμένα ωφέλη που τους δίνονται μέσω εμπορίου. Θέλουμε βέβαια να συνεχίσουμε να συζητάμε τα θέματα αυτά με την Επιτροπή σας και σε συνέχεια της, ε, του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο, που ε, είναι αρμόδιο ο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Όπω είπε και ο εισηγητής πολύ σωστά, θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέπεια μεταξύ του σχεδίου ψηφίσματο που συζητάτε αυτή τη στιγμή και του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ ε, στι Συμφωνίε εμπορίου. Όσον αφορά τώρα το θέμα της εταιρική κοινωνική Ευθύνη, να σας πω ότι επειδή αναφέρθηκε και από τον εισηγητή και από τον κύριο Σούλτς, Σαφώ δραστηριοποιηθήκαμε στο να υπάρχουν διάφανοι κανόνε ε, και σε διεθνέ επίπεδο, αλλά το εφελτήριο θα πρέπει να είναι μια εθελοντική εταιρική κοινωνική ευθύνη, διότι πηγαίνει πέραν των όσων απαιτούνται από νομική σκοπιά. Αυτό το οποίο εξετάζουμε και περιμένουμε με ανυπομονησία να το συζητήσουμε και με το Κοινοβούλιο, έχουμε συνεργαστεί και σε αρκετέ άλλε επιτροπέ του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, κυρίω ε, με την Επιτροπή απασχόληση να βεβαιωθούμε ότι όσοι κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη πραγματικά την υλοποιούν. Θα πρέπει όμως να ξεκινάμε επί εθελούσιας βάσης, διότι αλλιώς ε, είναι σαν να κάνουμε υποχρεωτικό κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, να ξαναδώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Oui, Monsieur le Président. ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι στη συζήτηση τα δύο βασικά ερωτήματα τα οποία έθεσα, του εθελοντικού υποχρεωτικού χαρακτήρα, είναι ένα από τα δύο ουσιαστικά ερωτήματα και το δεύτερο ερώτημα είναι το θέμα των κυρώσεων. Εγώ αναρωτήθηκα αν πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στις κυρώσεις, αλλά φαντάζομαι θα το διεξέλνουν το θέμα αυτό οι συνάδελφοι στις τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προθεσμία για τροπολογίες 16 Φεβρουαρίου. Όχι. Όχι. 14 Φεβρουαρίου. Σα 14 Φεβρουαρίου 6 η ώρα το απόγευμα. Πάμε στο σημείο 6. Ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και ανάπτυξη. Σχέδιο γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών. Πού είναι η αρμόδια για το θέμα αυτό. Ο εισηγητής μας είναι ο κ. Ζωζεφ Αντρές από τους Σοσιαλιστές αλλά και Δημοκράτες. Της δίνω μέσα στο λόγο. Σας δίνω το λόγο. Το κοπήραμε για το γεγονό ότι. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και τη συνεργασία με τον εισηγητή της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς και φυσικά η εδραίωση της ενιαίας αγοράς είναι μία από τις βασικές ε, από τους βασικούς θεμέλιους λήθους της στρατηγικής Ευρώπης 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για την οικονομική ανάπτυξη και η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους στόχους της ανάπτυξης, της εξάλληψης, της ένδυας και της επίτευξης των στόχων της χιλιετίας. Έχουμε θέσει στην έκθεση αυτή ερωτήματα τα οποία <clears throat> προφανώς συζητήθηκαν και πριν από λίγο. Το πρώτο ερώτημα που θέτουμε είναι ο αντίκτυπος που πρέπει να διακριβώνεται. Δηλαδή να υπάρχει ο έλεγχος του θετικού αντικτύπου για τις συμφωνίες και να βλέπουμε αν πρέπει να τροποποιηθούν οι ρήτρε όταν έρχεται για ανανέωση μια συμφωνία. Επίση, η ρήτρα κοινωνική εταιρική ευθύνη για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που μόλι συζητήσαμε, αν πρέπει να είναι δεσμευτική ή όχι. Εμεί σίγουρα θεωρούμε ότι πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε τροπολογία η οποία μπορεί να κατατεθεί, αλλά <clears throat> είναι γεγονό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ευθύνη για τα κοινωνικά θέματα και τα περιβαλλοντικά θέματα που μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι πρέπει οι εταιρείε να δεσμεύονται για την εταιρική ευθύνη. Πρέπει να μιλήσουμε για την ανταγωνιστικότητα τη ενιαίας αγορά και την ανταγωνιστικότητα ω βάση ανάπτυξη, αλλά μιλάμε για μια <clears throat> υπεύθυνη ανάπτυξη και από την πλευρά των επιχειρήσεών μας και την μη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μαϊμουδική παραγωγή ε, πειρατική ή μαϊμουδική παραγωγή και επίσης υπερεκμετάλλευση φτηνών εργατικών χειρών που μπορούν να οδηγήσουν σε μεταναστευτικές ροές και πολλά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι σημαντικό να, πει, να προπαροτρύνουμε τις εταιρείες, επιχειρήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να λειτουργήσουν στο παγκόσμιο αυτό στερέωμα, κάτι το οποίο πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν ανέφικτο συμφωνίες με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία ή η Βραζιλία είναι πολύ δύσκολες σε διοικητικό επίπεδο για να μπορέσουν να συμμετέχουν εταιρείε παραγωγικά σε δημόσιους διαγωνισμούς μέσα στα πλαίσια μιας διαφάνειας. Ο στόχος αυτής της ε, έκθεσης λοιπόν έχει σαν στόχο να τονίσει διάφορες πτυχές του διεθνούς εμπορίου, συγκεκριμένα την κοινωνική πτυχή που πολλές φορές δεν την αντιμετωπίζουμε επαρκώς, ώστε σε κάθε συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα να, είναι και μια κοινωνική, να υπάρχει και μια κοινωνική πτυχή που έχει να κάνει με την αλληλοβοήθεια στα θέματα αυτά. Εγώ φυσικά θα λάβω υπόψη τι απόψει οι οποίε θα διατυπωθούν και τι τροπολογίε οι οποίε θα κατατεθούν από του βουλευτέ τη Επιτροπή μα εν καιρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αρχίζει ο γύρος των ερωτήσεων πρώτο πρώτο τον κύριο Γιακολίνο που είναι και σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα μόλις ακούσαμε από τη συνάδελφο Βαρέα. Συμφωνώ με τις περισσότερες εξ αυτών. Θα πρέπει να άρουμε όλες τις συγκεκριμένες δυσκολίες, να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες ε, και να κάνουμε την ενιαία αγορά πραγματικά ανταγωνιστική. Συμφωνώ για τις παραγράφους που αναφέρονται στις κοινωνικές πτυχές. Βέβαια αναφερόμαστε στην ε, βιώσιμη και ευφυή ανάπτυξη. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε ίσως να ενισχύσουμε και την ενιαία αγορά των επιχειρήσεων, όπως επίσης θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε ότι αντί για την αντιμετώπιση του ντάμπινγκ μπορούμε να προβλέψουμε λίγο γενικότερα τι γίνεται με την παραβίαση των ε, διεθνών προδιαγραφών Θα πρέπει να αναφερόμαστε βέβαια στις καταχρήσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προτάσεις ε, ως προς την ανάγκη να άρουμε όλα τα προσκόμματα που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε ελεύθερη αγορά. θα υπάρξουν τροπολογίες από πλευράς μου. Ε, θεωρώ ότι από κάποιες από αυτές τις τροπολογίες θα μπορούσαμε ίσως να καταλήξουμε σε κάποιον ισορροπημένο συμβιβασμό με την εισηγήτρια, την οποία ευχαριστώ για την ευγενική ε, και πολύ ακριβή παρουσίαση που μας έκανε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Στέλλερ από τις Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης έχει καλές προθέσεις. Κάπου όμως έχουμε χάσει το στόχο και τη σαφήνεια. Δεν είναι σαφές, για παράδειγμα, τι εννοούμε όταν μιλάμε για ψηλέ προδιαγραφές ε, στην έκθεση. Μιλάμε για παγκόσμιες προδιαγραφές ή προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο αναφέρεται στην ενία αγορά που υποδηλώνει ότι μιλάμε για τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είχαν πρόβλημα οι πράσινοι με αυτό, αλλά αναφερόμαστε και σε πολυμερείς οργανισμούς που υποδηλώνει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει ίσως να είναι λίγο πιο σαφές το κείμενο σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ επίσης και με τους προλαλήσαντες. Υπάρχει ανάγκη να ε, συνδέσουμε τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ε, τα στάνταρ για το CSR με τις ε, παραβιάσεις. Ένας εθελοντικός κανονισμός, κανονικός, εθελοντικός κώδικος δεν έχει αποτέλεσμα. Το έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως. Δεν υπάρχει καμία επίκριση ουσιαστικά για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο, για την ανάπτυξη και τις παγκόσμιες υποθέσεις. Κάποιο είπε ότι υπάρχει συνοχή με την στρατηγική του 2020 εσωτερικός και το έγγραφο για το εμπόριο και τις παγκόσμιες υποθέσεις. Το ένα θα έπρεπε να είναι εξωτερική διάσταση του άλλου. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται αυτή τη στιγμή ε, αναφέρεται περισσότερο στις συνολικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι την ευφυή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020. Το σχέδιο γνωμοδότησης υποστηρίζει και την ε, προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Έχει γίνει όμως ουσιαστική συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας για τη ΣΑΚΤΑ και αυτά δεν αντικατοπτρίζονται, αυτά που συζητήσαμε δεν αντικατοπτρίζονται στο κείμενό σας. Θα παρουσιάσουμε τροπολογίες από πλευράς των Πρασίνων για όλα αυτά τα θέματα. Και εμείς φυσικά θα τα εξετάσουμε, ο Πρόεδρος. Πάντοτε εμπνέομαι από την Προεδρία σας κύριε Πρόεδρε μου. Γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Ναι, θα καταθέσουμε τροπολογίες στις 50 αυτές προτάσεις όπως θα το επιτρέψει ο χρόνος που διαθέτει το προσωπικό μας. Τώρα έχω πολλά να πω εδώ, αλλά επειδή είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα περιοριστώ μόνο στις πρώτες 25 προτάσεις. Θα είμαι λέει συντομότατος. Πρώτη πρόταση. Μιλάει για έναν εθνικό νόμο ευρεσιτεχνιών. Νομίζω ότι αυτό πράγματι θα ήταν πιο αποτελεσματικό από οτιδήποτε ενωσιακότερο. Δύο, ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Μα αυτό το ακούμε από το 60. Έχουμε ενιαία αγορά υπηρεσιών και αγαθών ή όχι. Το θέμα είναι ότι για τις υπηρεσίες ειδικά δεν έχουμε. Και για να τυποποιηθούν τα προϊόντα, αυτό που προτείνει η Ένωση, δηλαδή αντί να τυποποιηθούν τα προϊόντα, καλύτερα τα υπάρχοντα να μπορούν να πολλούνται σε ολόκληρη την Ένωση. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην περίπτωση Κασέλ της Διζών. Να απαντήσει η Επιτροπή. 11. Πρόταση 11. Μιλάτε για σχέδιο ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό ας το αφήσετε στο μηχανισμό καθορισμού των τιμών. Ενδιαφέρον όμως. 12, 13 και 14 υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι 15 ουδέτεροι, οι 16 και 17 εμποδίζουν απ' την άλλη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 17 προσέξτε πώς τελειώνει λέει να μπορούν οι δημόσιες συμβάσεις να υποστηρίζουν καλύτερα άλλα προγράμματα. Τι προτιμούμε λοιπόν, αποτελεσματικότερες συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών ή ή αγαθά και υπηρεσίες που να καθορίζονται κατά την παραγωγή τους από τις πολιτικές απόψεις κάποιου υπαλλήλου. 90. Λέει θα υπάρξει οδηγία για κοινή και κοινό και συνδυασμένο επιχειρησιακό φόρο. Θα υπάρξει δηλαδή ομοιομορφία στη φορολόγηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ένωση. Εδώ το θέμα είναι ότι ορισμένες πιο καθυστερημένες χώρες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο επιχειρησιακό φόρο από άλλες ή από η Γερμανία. Αυτό δεν το αναγνωρίζει η Κομισιόν και θα ήθελα να μου απαντήσει. Πρόταση 20 μιλάει για νέα στρατηγική του ΦΠΑ το 11 και λέει το 12% τη ΦΠΑ δεν συλλέγεται για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και τις πτωχεύσεις. Τι μας λέει εδώ η Κομισιόν, ότι οι εξαιρέσεις που αφορούν τις πτωχεύσεις θα καταργηθούν. Γιατί έτσι φαίνεται να εννοεί. Αφού υπάρχουν διαφορετικά ύψη ΦΠΑ στην Ένωση, τα οποία καθορίζουν οι εθνικές κυβερνήσεις, που δεν είναι βέβαια πάντα αλάθητες, ιδιαίτερα η κυβέρνηση του ΙΤΑΒ που έχει βάλει για ορισμένα αγαθά 20%, πώς μπορεί να πιστεύει η Κομισιόν ότι θα καθορίσει εκείνη καλύτερα και πιο αποτελεσματικά αυτό το ύψος. Και τώρα οι 25, τις επόμενες 25 θα τις ζητήσω την άλλη φορά. Οι 25 λοιπόν λέει ότι θα κάνει σχετική ανακοίνωση για τις υπηρεσίες κοινού, ε, γενικού συμφέροντος, αλλά γιατί δεν μας έχει ακόμη απαντήσει μέχρι τώρα στις απορίες των πολιτών και επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας μέχρι τώρα. Πολλοί από εμάς ανησυχούν για τις υπηρεσίες αυτές, δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Θέλουμε αποτελεσματικότερες δημόσιες επιχειρήσεις με επιχορήγηση ή την παρεμπόδιση αυτών από τον ενωσιακό νόμο τονίσω ιδιαίτερα προς τους σοσιαλιστές και σοσιαλίστριες εδώ ότι το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι δημόσιες υπηρεσίες δηλαδή. Να μην ξανακάνει τα ίδια η Κομισιόν με τον προηγούμενη της πρόταση όπου δεν υπήρχε καμία συνέπεια. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Η Κομισιόν. Πώς, πώς λέγεστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Προ. Λέγομαι Πάμελα Μπρούντερ. Και είμαι στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. Θα προσπαθήσω χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς η ομιλήτρια. Να αρχίσω από την αρχή. Όχι. Από τη μέση. Θέλω να χαιρετήσω καταρχήν το σχέδιο γνωμοδότησης που τονίζει τις εξωτερικές πτυχές της εσωτερικής αγοράς και που με τρόπο πολύ θετικό συμπληρώνει το σχέδιο κ. Μπουζόη στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς από τη δική μας άποψη ο αγώνας κατά της πειρατείας και της παραποίησης είναι πολύ σημαντικός και επίσης η έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετρία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές προμηθειών είναι πολύ σημαντική. Γενικά το θέμα της πρόσβασης σε αγορές τρίτων χωρών. Τούτου λεχθέντος. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε και ο συνάδελφός μου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης για τα, η συναδελφός μου μάλλον, για τα θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το αν πρέπει να είναι δεσμευτική ή όχι αυτή η ρήτρα. Παραπέμπω σε αυτά που σας είπε, γιατί αυτή είναι η πάγια θέση της Κομισιόν προς το παρόν, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε προς μια υποχρεωτική ρήτρα εταιρικής ευθύνης. Καταγράφω όμως τις δικές σας θέσεις και ανησυχίες. Και τώρα για τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν <clears throat> από τον τελευταίο ομιλητή. Προσπαθώ να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά. Για τα θέματα ευρεσιτεχνιών. Σας υπενθυμίζω ότι προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε διευρυμένη συνεργασία για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας. Η Κομισιόν έχει συλλέξει πολλά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι για να μπορούμε να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα είναι πρόσφορο για την καινοτομία και επανέρχομαι στη συζήτηση που είχατε προηγουμένω για την Ένωση της Καινοτομίας είναι σαφές για την Κομισιόν ότι το να μπορεί να υπάρχει προστασία των ευρεσιτεχνιών στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγον για την ενωσιακή ανταγωνιστικότητα, ιδίω για τις μικρές αλλά και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι πιο φτηνό αυτό το σύστημα από αυτό που επικρατεί τώρα και επομένω θεωρούμε ότι είναι μια κέρια προτεραιότητα και αυτό δεν έχει τύχει διαφυσβήτηση ούτε από τα κράτη-μέλη πέραν αυτών βέβαια που δεν μπορέσανε να συμφωνήσουν στην συμβαστική λύση η οποία παρουσιάστηκε υπό τη υποβελική προεδρία. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι πολύ πιστικό αυτό το, για να δείξει τι μπορούμε να κάνουμε νομοθετικά για να προωθήσουμε την καινοτομία. Δεύτερον, η ενιαία αγορά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε σχέση με την υπόθεση Cassis de Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μια οδηγία για τις υπηρεσίες η οποία συζητήθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο <clears throat> και τώρα τίθεται σε εφαρμογή και γι' αυτό εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή της από τα κράτη-μέρη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σε τελική ανάλυση να καταλήξουμε σε μια κοινή αγορά υπηρεσιών. Επίσης είναι σαφές ότι η ισορροπία μεταξύ μιας αποτελεσματικής πολιτικής προμηθειών όπου οι εθνικές αρχές θα διαλέγουν την καλύτερη τιμή και την καλύτερη, το καλύτερο επίπεδο παροχών που σημαίνει να προωθήσουμε και πράσινα προϊόντα, να εξασφαλίσουμε κοινωνικές υπηρεσίες και την καλύτερη ποιότητα, να το εξισορροπήσουμε αυτό με το θέμα της αμοιβαιότητας στους δημόσιου διαγωνισμούς. Να τα εξισορροπήσουμε και όχι να τα θέσουμε σε μετοπική σύγκρουση όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να θέσουμε να αφιβόλο την αποτελεσματικότητα των δημοσίων διαγωνισμών για την αμοιβαιότητα. Για τα θέματα της φορολογίας, ούτε στα θέματα του ΦΠΑ, ούτε σε εταιρικό φόρο, θα προτείνει η Κομισιόν μια συγκεκριμένη εναρμόνιση και η Κομισιόν παρόλα αυτά θα έλθει ταχαίως με προτάσεις και με μια έκθεση αξιολογήσεως αντικτύπου σε σχέση με την εδρεωμένη εταιρική βάση φορολογήσεως για επιχειρήσεις που θα καταδείξει ποιο είναι το κόστος των επιχειρήσεων μέσα στην ενία αγορά. Τέλος για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, αυτό το οποίο κάνουμε στον τομέα των δημοσίων προμηθειών επίσης, είναι να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε <clears throat> υπάρχει πλήρης ελευθερία στην ε, αρχή η οποία είναι αρμόδια για τους δημόσιους διαγωνισμούς ώστε να δράσει με τρόπο ευέλικτο και να έχει την απαραίτητη ελευθερία επιλογής για το αν θέλουν να κρατήσουν κάποιες υπηρεσίες μέσα στο δημόσιο χώρο ή να τις δώσουν σε ιδιωτικούς φορείς. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να τρέφεται οποιουσδήποτε φόβους για τα μελλοντικά σχέδια της Κομισιόν τα πράγματα πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προτού δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Σαζάλ να με αντικαταστήσει γιατί πρέπει να φύγω για λίγο. Μπορείτε να θέλετε να με αντικαταστήσετε. Ζωζέφα, έχει το λόγο. Eh, eh, gracias, presidente. Eh, como estaba usted preguntando, no sabía lo que quería. Όταν ε, θέσετε την ερώτηση δεν είχα καταλάβει σε τι απευθύνεστε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ του πάντε για τη συνεισφορά τους. Ε, κατάλαβα ότι ο καθένα θέλει να αφήσει το σημάδι του ανάλογα με την πολιτική ομάδα που εκπροσωπεί. Προφανώ εγώ ανήκω στη σοσιαλιστική ομάδα και θα ήθελα να υπάρχει κοινωνικό χαρακτήρα ε, στις εμπειρικές συμφωνίες. Είναι ε, γνωμοδότηση ε, προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ που είναι η αρμόδια επί της Επομένως δεν μπορώ να επεκταθώ πάρα πολύ. Υπάρχει περιορισμό στον αριθμό των χαρακτήρων ε, στις γνωμοδοτήσεις αυτές και προσπάθησα να επισημάνω τα πιο σημαντικά. Ο κοινωνικός χαρακτήρας για την ομάδα των σοσιαλιστών είναι ζωτική σημασία φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν πραγματικές επικρίσεις, ε, διότι πρόκειται για μία γνωμοδότηση και δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε για ένα θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τροπολογίες που μπορεί να βελτιώσουν το, την κατάσταση. Ε, και για τον εισηγητή που έκανε μια πιο γενικευμένη κριτική, να πω ότι η ενιαία αγορά είναι μία διέξοδος για να ε, διαφύγουμε από την κρίση δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ότι είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας και δεν βελτιώνει τις επιχειρήσεις. Ίσα ίσα θεωρούμε ότι βοηθά τις επιχειρήσεις να ξεφύγουν από την κρίση μέσω της ενιαίας αγοράς. Είμαι ε, στη διάθεσή σας ε, για προτάσεις ε, και συμβουλές, να προσπαθήσω να βελτιώσω όσο το δυνατόν καλύτερα το κείμενο, γιατί στο τέλος, τέλος αυτό επιθυμούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω τις προθεσμίες για τις τροπολογίες 14 Φεβρουαρίου. Είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και τώρα περνάμε στο σημείο 7 της διάταξεις. διάταξης. Συμφωνία εταιρική σχέσης καθώς και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ. Ο συνάδελφός μας Εμίλιο Μενέντες Δεβάγε είναι ο εισηγητή για το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εμίλια, εάν θέλει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, φύγει ο Πρόεδρος Μορέιρα και σας ε, δώσει εσάς τη σκητάλη της Προεδρίας, που είστε εξίσου αποτελεσματικός, ήθελα να πω ότι ο Πρόεδρος Μορέιρα αποτελεί έμπνευση για όλους, όχι μόνο για τον συνάδελφο Ντάρτμουθ. Θα το λέω αυτό γιατί θα κάνω μία απόπειρα να δω κατά πόσο μπορώ να τραβήξω την προσοχή σας ε, για το κείμενο που θα σας παρουσιάσω. Δεν θα ήταν παράτολμο να πω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική γνωμοδότηση της ΣΥΝΤΑ. Ε, το περιεχόμενό της είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αναφερόμαστε στην κατάσταση μιας χώρας ε, όπως είναι το Ιράκ που έζησε όλα αυτά που έζησε και τα γνωρίζετε όλοι. Δεν θα επεκταθώ τώρα στα του Ιράκ. Να πω μόνο ότι για να υπάρχει επιτυχή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ σε πολιτικό και εμπορικό επίπεδο χρειάζεται σταθερότητα στη χώρα διότι χωρίς σταθερότητα, και αυτό είναι και το θεμελιώδες, δεν θα υπάρχει πραγματικό εμπόριο, δεν θα υπάρχουν επενδύσεις και θα βαλτώσει η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ιράκ. Για να μην σα κουράσω, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια σύνεοψη αυτών που έχω ετοιμάσει. Θεωρώ ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ κινούνται ταχύτατα σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν πριν από κάποια χρόνια, που όπως γνωρίζετε η μόνη παρουσία ε, που είχαμε μετά από την εισβολή στο Ιράκ του 2003, η μοναδική σημαντική περιουσία ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αρχίζουν να αλλάζουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο μερών και κινούνται πλέον σε τρεις πυλώνες. Ε, καταρχάς η σχέση σύνδεσης και συνεργασίας που συζητάμε και σχολιάζουμε, Δεύτερον, υπάρχει το μνημόνιο συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ, που αναφέρεται σε ενεργειακά θέματα. Και τρίτον, ο τρίτος πυλώνας, η χρηματοοικονομική βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία και αν δεν κάνω λάθος, από το 2003 ε, έχουμε δώσει ένα δις ευρώ. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η σχέση σύνδεσης και συνεργασίας είναι ο πρώτος σημαντικός σύνδεσμος που θα έχουμε μεταξύ των δύο μερών. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό νομικό πλαίσιο και για τις πολιτικές αλλά και για τις εμπορικές υποθέσεις. Γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2006, ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2009 και τώρα βρισκόμαστε πλέον εν αναμονή της κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, υποθέτουμε ότι θα γίνει εντό του έτου. Υποθέτουμε τουλάχιστον. να σας πω ποια θεωρώ ότι είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Καταρχάς, πριν από την εμπορική πτυχή και δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς δεδομένης και της κατάστασης του Ιράκ, υπάρχει ο πολιτικός διάλογος και ο διάλογος ασφαλείας με το Ιράκ σε όλες τις συμφωνίες αυτής της μορφής, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να υπάρχουν πάντα και υπάρχουν οι διάσημες ρήτρε ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Αυτό είναι απαραίτητο και πρέπει να υπάρχει. Στην συμφωνία έχουμε σοβαρή αντιμετώπιση των θεμάτων ενέργειας, επενδύσεων, ε, περιβάλλον, δικαιοσύνη κλπ. κλπ. Αλλά επίσης καθορίζονται και κάποιοι μηχανισμοί ώστε να υπάρχει σωστή υλοποίηση και εφαρμογή της συμφωνίας. Δύο λόγια τώρα για τις εμπορικές πτυχές. Γνωρίζετε ότι το Ιράκ δεν ανήκει στον ΠΟΕ, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς άλλωστε. Η Ευρώπη βέβαια εκτιμά ότι παρά το γεγονός ότι το Ιράκ δεν ανήκει στον ΠΟΕ, η συμφωνία διέπεται από τους κανόνες, ε, τη φιλοσοφία και τις μεθόδους που ακολουθεί ο ΠΟΕ. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώ. Εάν θέλουμε το Ιράκ ε, σταδιακά να προοδεύσει και να περάσει στην πλήρη ένταξή του στη διεθνή κοινότητα και στη διεθνή οικονομία και στις παγκόσμιες αγορές. Δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή από αυτή που προτείνει ο ΠΟΕ για αυτή την περίπτωση. Έχει προβλεφθεί επίσης ε, και ένας κατάλληλος μηχανισμός για επίλυση διαφορών και δεδομένων των συνθήκων είναι πολύ σημαντικός αυτός ο μηχανισμός, γι' αυτό άλλωστε και συμπεριλαμβάνεται και στο, στη συμφωνία. Υπάρχουν και κάποιες πτυχές που αναφέρονται στις ε, δημόσιες αγορές, στις επενδύσεις και στις υπηρεσίες. Τέλος, ε, ε, ολοκληρώνοντας, να σας ε, πω δύο λόγια για τους βασικούς στόχους αυτής της συμφωνίας. Όπως σας είπα καταρχάς, κυρίως η σταθερότητα. Πρωτίστως η σταθερότητα, διότι χωρίς τη σταθερότητα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αυθεντικού εμπορίου και επενδύσεων ε, ουδεμίας μορφής. Στη συμφωνία Επίσης ε, προάγονται και προωθούνται οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ευτυχώς ήδη έχουν ξεκινήσει στο Ιράκ. Μπορεί να ακουστεί ε, και ως κάτι το οποίο λέμε επανειλημμένος, αλλά ε, δεν αρκεί να το πούμε όσο περισσότερες φορές γίνεται, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τους Ιρακινούς, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και εμπόριο από σε διμερές επίπεδο ε, και όπως σας είπα ε, τηρούνται οι κανόνες του ΠΟΕ παρά το γεγονός ότι το Ιράκ δεν ανήκει ακόμα στον ΠΟΕ. Επειδή είναι αυτή της μορφής η συμφωνία και επειδή πρόκειται για το Ιράκ, η νομική ασφάλεια και ε, στις διμερείς σχέσεις είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική επίσης και η διαφάνεια και να μην ε, υπάρχει συνεργασία και να φαίνεται ότι οι σχέσεις μας είναι σαν να είναι ο ένας από τον Άρη και ο άλλος από την Αφροδίτη. Ε, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι στην καθημερινότητά μας και θα αναφέρεται στις καθημερινές συναλλαγές μας και επενδύσεις. Εν κατακλείδη, το θέμα του Μνημονίου Συνεννόησης για την Ενέργεια, να σας πω ότι πρόκειται για ένα μέσο το οποίο μας επιτρέπει... Ε, επειδή ακριβώς έχει και πολύ μεγάλη πολιτική βαρύτητα, ε, δεν έχουμε όμως ακόμα την κατάλληλη νομική βαρότητα. Αυτό θα γίνει μόλις κυρωθεί η συμφωνία σύνδεσης και συνεργασίας που συζητάμε. Ελπίζω να μην ακρηγόρησα. Θα σταματήσω εδώ και περιμένω σχόλια από τους παριστάμενους ή δεν ξέρω αν έχει προεδρία κάτι άλλο να μου πει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους της Επιτροπής μας και στην Εκτελεστική Επιτροπή θέλω να υπογραμμίσω δύο πτυχές του θέματος αυτού όπως είπε ο συνάδελφος Μενένδες. Πρώτον, η συμφωνία αυτή περιέχει και μια εμπορική πτυχή που είναι φυσικά η πιο σημαντική. Αλλά μόλον τούτο η Επιτροπή μας βρίσκεται κάπως παριγκονισμένη στη συμφωνία αυτή για την εταιρική σχέση και ως ε, εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων, ως συντονιστές, έχουμε <clears throat> προσπαθήσει να αξιολογήσουμε καλύτερα το ρόλο που πρέπει να έχει η Επιτροπή μας σε τέτοιου είδους εταιρικές ε, σχέσεις συνεργασίας. Διότι δεδομένου του τεράστιου ειδικού βάρους του εμπορικού πυλώνα δεν είναι λογικό η δική μας Επιτροπή να συμμετέχει τόσο λίγο σε αυτή τη διαδικασία και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να θέσω και υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας σκεφτεί λιγάκι για το θέμα αυτό είναι πώς βλέπει η Κομισιόν το ρόλο του Κοινοβουλίου μέσα στο πλαίσιο αυτό η εντύπωση που σχημάτισα εγώ είναι ότι <clears throat> εφόσον έχουμε για μια συμφωνία Trade and Partnership Agreement, μια συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα και εμπορική όμως, ίσως θα πρέπει η Επιτροπή ΙΝΤΑ να αναλάβει ένα πιο σημαντικό ρόλο, γιατί ουσιαστικά έχουμε τη μεγάλη ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αξιολόγηση αυτών των συμφωνιών. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν, όπως θα θέλαμε και από την Κομισιόν, θα εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε η Επιτροπή μας να παίξει πλήρως τον ρόλο της σε αυτού του είδους τις συμφωνίες. <clears throat> Νομίζω ότι αυτό είναι η σωστή κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και τώρα ζητώ στους συναδέλφους εάν θέλουν να λάβουν τον λόγο. Ο κύριος Τέιλο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η παρέμβαση, η εισαγωγική παρέμβαση του κυρίου Μενέντες. Ο κύριος Μενέντες τόνισε την επιζήτηση σταθερότητας που είναι στο Ιράκ, που είναι φυσικά μια, ένα προαπαιτούμενο και εμείς ανησυχούμε πολύ για το γεγονός ότι η σταθερότητα στο Ιράκ κινδυνεύει να υποσκαφθεί από μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή ελάχιστα ελέγχει τη χώρα αυτή και έχει πολύ μικρή νομιμοποίηση ούτε ξέρουμε αν έχει την ικανότητα να διαπραγματευτεί μία διεθνή <clears throat> συνθήκη αυτόνομα ως κυβέρνηση. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη συζήτηση που πρέπει να διεξαγάγουμε. Και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και εσάς από τη δική σας οπτική γωνία αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Και με την ευκαιρία αυτή να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι οι Ιρακινές αρχές ξέρουν τι θα παραδώσουν με την υπογραφή τους για, τις, ε, ε, για τους εθνικούς πόρους και τις επενδύσεις σε σχέση με το ανώτατο όριο για τη ε, συμμετοχή από ξένους στις επιχειρήσεις τους, τα θέματα μεταλαμβάνευσης τεχνολογίας, τα θέματα ευθύνης των επενδυτών να καθαρίσουν το περιβάλλον μεσαϊσαγωγικά, εισαγωγικά προτού φύγουν από τη χώρα τους. Γιατί είναι σαφέ ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μονάχα οικονομικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα παγκόσμια σταθερότητα και τοπικής οικοδόμησης τη ειρήνης. Και για το λαό του Ιράκ θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο περιθώριο μέσα στις οικονομικές πολιτικές που ακολουθηθούν για να επιτευχθούν και αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Καμπέλ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να ρωτήσω δύο πράγματα το ότι κινούμαστε προς μία τέτοια συμφωνία με το Ιράκ σημαίνει ότι αναγνωρίζει πολιτικά η Ένωση τη νέα κυβέρνηση του Ιράκ ή όχι. Μετά τον πόλεμο εκεί τίθεται το ερώτημα. Δεύτερον, είχε υποθεί ότι οι δύο μεγαλύτεροι πιστωτές του Σαντάμ ήταν οι Ρώσοι και οι Γάλλοι οι οποίοι όμως αντιτάχθηκαν και οι δύο στον πόλεμο και αυτή τη στιγμή θεωρείται αξιόπιστο το Ιράκ ότι μπορεί να αποπληρώσει δηλαδή τα χρέη που είχε δημιουργήσει με αυτές τις δύο χώρες. Μπορεί να υπάρχει συμφωνία με μια χώρα αν δεν είναι αξιόπιστη αξιόχρεη. Ο Δανιήλ. Συζητούμε τώρα την ε, εμπορική μας σχέση με το Ιράκ στο μέλλον. Και το θέμα αυτό έχει ήδη αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή μας στο παρελθόν, στην προηγούμενη θητεία. Θα ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν αν εξασφαλίσει με, τα, με τις προτάσεις να καταλήξουμε, ότι θα καταλήξουμε σε μια διαφοροποιημένη οικονομία στο Ιράκ με ποικίλε δραστηριότητε. Θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν τι προτείνει για να μπορεί η οικονομία του Ιράκ να μην βασίζεται 100% στις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά να έχει και άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες. Και πώς αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη ευμάρεια των πολιτών του Ιράκ. <clears throat> Εντάξει. Η Κομισιόν, ο κύριος Ολιβιέ Ντελαροσίλα, πληρέστατος ήταν για τα θέματα αυτά. Περιορίζω τον εαυτό μου να κάνω μερικές παρατηρήσεις μονάχα και να προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία άπτονται άμεσα τη συμφωνίας αυτής. Ο στόχος της συμφωνίας ήταν, όπως είπατε, να εξασφαλίσουμε ένα νομικό πλαίσιο που δεν θεσπίζει διακρίσεις και το οποίο έχει σταθερότητα για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις στο Ιράκ και επίσης να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και τους βασικούς κανόνες του ΠΟΕ στη συμφωνία αυτή, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα των συναλλαγών, αλλά και την μελλοντική δυνατότητα προσχώρησης στο ΠΟΕ. Κάτι το οποίο δέχτηκαν οι Ιρακινοί, διότι ενσωμάτωσαν τις βασικές αρχές του ΠΟΕ, που είναι πολύ σημαντικές. Όπως η ρήτρα του πλέον ευνοουμένου έθνους, το σύστημα <clears throat> αξιολόγησης για τα τελωνία, την ε, μείωση των ποσοτικών προπεριορισμών που είναι βασικά στοιχεία της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το παραγνωρίσουμε, είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα τη στιγμή που έχουμε μια αρνητική στάση της Λιβύης ως παράδειγμα. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό τώρα να κατανοήσουμε το εξή. Εμεί χρειάστηκε στη μέση του δρόμου να τροποποιήσουμε την προσέγγιση μα στι διαπραγματεύσει, γιατί οι Ιρακινοί, παρά την θέλησή του <clears throat> να περατωθεί αυτή η συμφωνία, δεν είχαν ούτε την απαραίτητη νομοθεσία, ούτε το τελωνιακό σύστημα, ούτε νομοθεσία για την πνευματική κτησία, ούτε για τις δημόσιες προμήθειες και δεν είχαν και την διοικητική ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Δείξαμε μεγάλη ευκαμψία λοιπόν, μειώσαμε τις φιλοδοξίες μας, προβλέψαμε να υπάρχουν ερήτερες συνάντησεις στο μέλλον και ορισμένες ρυθμίσεις ad hoc. Αυτό <clears throat> σημαίνει ότι αποδεθήκαμε σε ένα θετικό εγχείρημα, διότι και ένας άλλος στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να ανοίξουν οι αγορές του Ιράκ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, να υπάρχουν προϋποθέσεις για συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς και εκεί έχουμε ένα συγκεκριμένο κεκτημένο που οι Ιρακινοί δεσμεύονται να το συνεχίσουν. Για την παροχή υπηρεσιών υπάρχει μια ρήτρα διαφύλαξης που επιτρέπει στο βαθμό που αναπτύσσεται η νομοθεσία τους να προσαρμοστούν οι δεσμεύσεις τους. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα το οποίο θέσατε, στα ερωτήματα καλύτερα, η διαφοροποίηση της οικονομίας του Ιράκ. Όπως σε όλες αυτές τις συμφωνίες, η διαφοροποίηση οικονομίας είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. <clears throat> Έχουμε μια συμφωνία πλαίσιο που προβλέπει συνολικές συνθήκες ώστε να μπορέσουν οι εθνικοί φορείς και οι ευρωπαϊκοί φορείς να συμμετέχουν σε μια διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας με αποτελέσματα τα οποία θα εξαρτηθούν φυσικά από την εσωτερική εφαρμογή πολιτικών προς την κατεύθυνση αυτή. Είδαμε στο παρελθόν με την Αλγερία ότι ήταν μέτριο το αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία πλαίσιο που δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ιρακινό νομοθέτη ή τον χαράκτη εθνικής πολιτικής. Μπορούμε να συνάψουμε τώρα συμφωνίες με μια χώρα για την οποία πλανώνται αμφιβολίες για την φερεγγιότητά της. Εδώ έχουμε και τη συμφωνία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες θα κατασταθούν εκεί, οι οποίες θα απολαμβάνουν τον ίδιο συνδικών με τις εγχώριες εταιρείες. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι και μια εγγύηση μη διακρίσεως ότι θα έχουν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν προς το παρόν για τα ερωτήματα αυτά τα οποία απευθύνθησαν στην εμπορική διάσταση για τα θέματα της εταιρική σχέσης. Εδώ δεν θέλω να επισέλθω στη συζήτηση για το ρόλο του Κοινοβουλίου στην έγκριση αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι το στοιχείο της εταιρική σχέσης προεκρίθη από τους διαπραγματευτές για να τονίσει το γεγονός ότι έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία από ό,τι προβλεπόταν στο, στην αρχή. Προχώρησε λοιπόν θετικά αυτή η διαπραγμάτευση και θέλουμε να τονίσουμε τον ρόλο της αναγνώρισης προς το Ιράκ, δίνοντας στη συμφωνία ένα πιο ευρύ τίτλο από ό,τι προβλεπόταν καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μενένδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε σε κάποιες από τις ερωτήσεις και σε κάποια από τα σχόλια τα οποία έγιναν εδώ από κάποιους συναδέλφους. Δεν απάντησε, ίσως βέβαια δεν είναι και κατάλληλη στιγμή και δεν είναι και ο αρμόδιος, στην παρατήρηση του Πρόεδρου Ζαντό για την πιθανή συμμετοχή της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ στο θέμα αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίσουμε το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Επιτροπή μας. Να επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, ότι απαντήθηκαν κάποιες από τις ερωτήσεις και κάποιες από τις παρατηρήσεις σας, αλλά δεν ε, είπε τίποτα από αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, την, ε, το γεγονός ότι παραγωνίζεται την Επιτροπή μας ε, και το γεγονός ότι πρέπει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο η Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πρέπει να μας απαντήσετε κάτι. Να πω στον συνάδελφο Τέιλορ ότι εγώ θεωρώ ότι η Ιρακινή κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο δεν ελέγχει μεν τα πάντα, ούτε ή δεν τα ελέγχει επαρκώς, αλλά η συνομιλία γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας κυβέρνησης την οποία δεν θα σχολιάσω αυτή τη στιγμή ούτε την ομιμότητά της ούτε τον τρόπο που δρά. Δεν είναι εδώ ο τόπος να, να συζητηθεί αυτό. Είναι η κυβέρνηση με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτικές καταρχάς σχέσεις και με τη συμφωνία αυτή και εμπορικές σχέσεις ειλικρινά αγαπητέ συνάδελφε Τέιλορ, εγώ είμαι πιο αισιόδοξο από εσά. Θεωρώ ότι ε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε οι Ιρακινοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θα υπογράψουν. Έχουν και του κατάλληλου συμβούλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι ευρωβουλευτές ε, νομίζω μπορούν να εξετάσουν και αυτοί ε, και ξέρουν τι ακριβώ θα υπογράψουν. Στο συνάδελφο Κάμπελ τώρα Εγώ ξεκινώ από την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την κυβέρνηση, διότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με κάποιον εάν δεν υπάρχει ε, πολιτική της αναγνώριση και δεν υπάρχει διπλωματική αναγνώριση. Δεν ξέρω βέβαια να σας απαντήσω για το κατά πόσον επιστράφηκαν όλες οι πιστώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαρευνήσουμε. Δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή στον συνάδελφο Κάσπαρη. Νομίζω ότι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιον τρόπο, διότι εγώ δεν το ανέφερα πριν για να μην ε, μακρηγορήσω, αλλά το 99,9% των, επενδύσεων, των ε, εισαγωγών συγγνώμη, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ιράκ είναι πετρέλαιο. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι κατάλληλη αυτή η διαφοροποίηση. να πω ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άτυπη επίσημη συνάντηση και για τροπολογίες ε, για να έχουμε κάτι το οποίο δεν θα είναι απλώς ε, μία ανταλλαγή απόψεων αλλά να έχουμε ένα πιο ουσιαστικό κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Θα συζητήσουμε στους συντονιστές και συντονίστριες τον καλύτερο τρόπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα εταιρικής συμφωνίας. Ε, τώρα περνάμε στο σημείο οχατό. Σας υπενθυμίζω γιατί είναι το χρονοδιάγραμμα πολύ πεπιεσμένο. 3 Μαρτίου έγκριση και θα υπάρχουν μόνο 24 ώρες για την κατάσταση των προλογιών, 16 Μαρτίου στην Επιτροπή Ψηφοφορία. Το 8 λοιπόν τώρα η Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών μεταξύ Ένωσης και Καρέας. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε αναβάλει την ψηφοφορία όχι μόνο για τη ρήτρα ασφαλείας αλλά για όλο, όλη την έκθεση για σήμερα για να μπορέσουν λέει οι πολιτικές ομάδες να εξετάσουν δεόντως την πολιτική ως προς την Κορέα, τις κλιματολογικές αλλαγές για την πολιτική της ως προς αυτές, τις εκπομπές της διοξιδίου του άνθρακος, από αυτοκίνητα. Φαντάζομαι ότι κάθε ομάδα μπόρεσε να μελετήσει τα πράγματα και σήμερα θέλουμε να μας πει η Κομισιόν πώς αναλύει την πολιτική αυτή με την Κορέα ως προς την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος από τα αυτοκίνητα και γενικότερα όμως για την ε, Συμφωνία Ελευθερών Εναλλαγών μεταξύ, Εναλλαγών μεταξύ Ένωσης και Κορέας και μετά, μετά θα γίνει συζήτηση. Ο κύριος Γαρθία Μπερθέρο έχει πρώτο στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω βασικά να πω μόνο δύο πράγματα. Η Κομισιόν φυσικά χαιρετίζει την ψηφοφορία της ίντε για τη ρήτρα ασφαλείας. Ήταν πολύ σημαντικό. και πρώτη απόφαση της Επιτροπής σας υπό τη διαδικασία, σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης. Αναμένουμε σήμερα να δούμε τι θα πείτε γενικότερα για τη συμφωνία. Από ό,τι ξέρω, πριν ψηφίσετε θέλατε να σας πούμε, να σας κάνουμε μία αξιολόγηση γενικότερα. Δύο σημεία. Πρώτον, η νομοθεσία που πρόκειται να εγκρίνει η Κορέα σύντομα για τις εκπομπές και η συμπληρωματική συμφωνία της με τις Ηνωμένε Πολιτείες για τις ελεύθερες συνταλλαγές είναι τα θέματα που θα θίξω. Η νομοθεσία της Κορέας για το διοξίδιο του άνθρακος πρώτον. Κάναμε μία ενημέρωση όπου απαντήσαμε ερωτήσεις που έθεσαν οι Ευρωβουλευτέ και Ευρωβουλεύτριοι και αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις να μου τις θέσετε. Αλλά για μας δύο είναι τα σημαντικά θέματα που έχουν επιτευχθεί. Πρώτον, οι αλλαγές που ανακοίνωσε το Κορεατικό Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις εκπομπές διοξιδίου ανταποκρίνονται σε αυτά που είχαμε πει και εμείς και οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι ότι δηλαδή η αρχική πρόταση θα τους επιβάρυνε αδικαιολόγητα. Αυτό τώρα λύθηκε και η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος παίρνει υπόψη της όλα αυτά τα στοιχεία. Ήδη γραπτά σας δώσαμε πληροφορίες αν όμως θέλετε μπορώ να υπησέλθω και σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Το άλλο θέμα είναι ότι αυτά όλα γίνανε με τρόπο που δεν μείωσαν καθόλου τις υποσχέσεις που δέχτηκε η Κορέα να μειώσει τις εκπομπές της. Είχαμε, κάναμε συνομιλίες με τους εταίρους μας στην Κορέα και μας υποσχέθηκαν ότι δεν θα στρεβλώσουν το στόχο που είχαν ανακοινώσει για τις μειώσεις. Ελπίζω και στην τεχνική μας ενημέρωση να σας έχουμε δώσει επαρκείς διασφαλίσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η νομοθεσία που ανακοίνωσαν οι Κορεάτες λύνει τα προβλήματα αυτά και ότι επομένως δεν υπάρχει λόγος το Κοινοβούλιο να αμφισβητήσει και να μην εγκρίνει. Το δεύτερο θέμα είναι ότι, αν και δεν το είπαμε από την αρχή, είναι η συμπληρωματική συμφωνία της Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Δεκέμβριο για ορισμένες πτυχές της συμφωνίας τους ελευθέρων συναλλαγών. Ο Παύλος Σάλβα μα σας είχε δώσει ορισμένα στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η αξιολόγηση της Κομισιόν είναι ότι αυτή η συμπληρωματική συμφωνία με κανέναν τρόπο δεν αμφισβητεί την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαίων εξαγωγών στην κορεατική αγορά. Ιδιαίτερα αναφέρομαι σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει ηθική ήτρα ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά εκεί δεν λέγεται τίποτα που να διαφέρει από αυτά που λέμε και στις γενικές ρήτρες ασφαλείας που διαμαρτυρθήκαμε και εμείς με τους Κορεάτες. Τίποτα ιδιαίτερο λοιπόν που να αμφισβητεί ή να θέτει τους αυτοκινητοβιομηχάνους των Ηνωμένων Πολιτειών σε δυσμενέστερη θέση από τους Ευρωπαίους. Δεύτερον, έχουν ακουστεί ερωτήματα για τις εξαιρέσεις που θα ενέφερε η συμπληρωματική αυτή συμφωνία και πάλι δεν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εξαγωγή είναι σε δυσμενέστερη εξαγωγική θέση. Θα παρακολουθήσουμε βέβαια στενά και το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά και στην ομάδα εργασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία θα διασφαλίσουμε ότι η Κορέα θα πληρεί πλήρως όλα αυτά τα οποία έχει δεχτεί τέλος. Βεβαίως η Κομισιόν χαίρεται ιδιαίτερα για τη συνεργασία της με την Επιτροπή σας και ελπίζουμε σήμερα να ψηφίσετε θετικά και αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο είμαστε στη διάθεσή σας. ρηθούμε ο συνάδελφός μας Ροβέρτος που είναι μεγά, μέγας γνώστης της συμφωνίας αυτής και εισηγητής επομένως ήδη θέλει να μιλήσει ορίστε Ροβέρτο Ευχαριστώ Συγγνώμη καθυστέρησα λίγο αλλά στην Αγγλία κάθε φορά που έχει κακό καιρό και φυσάει δεν πετάνε τα αεροπλάνα, ενώ θα έπρεπε. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να πω ότι αυτά που μόλις είπατε, Γνάθιο, καταδεικνύουν ότι εργαστήκατε πολύ σκληρά. Εμά μα ανησυχούσαν πάντα οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Ήταν ένα θέμα για το οποίο δεν είχαμε επαρκείς πληροφορίε. Νομίζω ε, έγινε μια συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα και πολύ καλά την εξηγήσατε θεωρώ ότι είμαι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα πλέον. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια πολύ ξεκάθαρη υπόθεση μέσω του μηχανισμού διασφάλισης και το Πάμπλο Σάλβαρο καταφέραμε να επιλύσουμε το θέμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να βασιζόμαστε μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά το γεγονός ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έκαναν εξαιρετική δουλειά. Θεωρώ λοιπόν ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Δεν έχω κάποια περαιτέρω προβλήματα. Θέλω να προχωρήσει ψηφοφορία για να περάσει το θέμα. Για όσους δεν υπερψηφίσατε τη συμφωνία ε, ε, ελευθέρω εμπορία με την Κορέα, να σας πω τα εξή. Σήμερα το πρωί στις 6 το πρωί σε ένα από τα εθνικά δίκτυα ε, υπήρχε μια συζήτηση για τις εμπορικές συμφωνίες και υπήρχαν εμπειρογνώμονες που έλεγαν ε, ότι αυτή η συμφωνία εμπορίου είναι εξαιρετική, θα οδηγήσει σε ευημερία μαζί με όλες τις υπόλοιπε εταιρικέ ε, ε, σχέσεις εμπορίου θα οδηγήσει ευημερία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως για πρώτη φορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Βρετανία ε, μίλησαν για κάτι σωστά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τους σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση αυτή και ζητώ συγγνώμη για άλλη μια φορά για την καθυστέρησή μου. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Παύλο Σάλμπα Παύλο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βεθέρο και για τη δουλειά του και για όλες τις διευκρινήσεις που έκανε. Κατάφερε να επιλύσει αρκετά θέματα. Στη ε, διάρκεια της ψηφοφορίας της ρήτρα διασφάλισης ε, και εγώ και ο πρόεδρος και οι άλλοι συνάδελφοι εκτιμήσαμε τη βοήθειά σας και καταφέραμε να έχουμε ε, θετικό αποτέλεσμα και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που θα ψηφίσουμε τώρα. Από πλευράς μου έχουν διευκρινιστεί όλα τα θέματα. Για μένα είναι όλα σαφή και για τη συμφωνία για το διοξίδιο του άνθρακα και την ε, σχέση Κορέας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα θέμα μόνο που θα ήθελα να μου διευκρινίσετε. Εδώ και πέντε χρόνια, συγγνώμη, για πέντε χρόνια οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρέπει να προσαρμοστούν σε 29 προδιαγραφές, σε ένα κόστος το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό. Στη διάρκεια αυτών των πέντε ετών έγινε και διαπραγμάτευση για η κατασκευή 25.000 αυτοκινήτων στην Κορέα, τα οποία δεν πληρούν καμία από αυτές τις προδιαγραφές. Θα υπάρχει λοιπόν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτιο για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να μου το διευκρινίσετε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Merci σκιώδη συζητητέ οι οποίοι θα θέλαμε να λάβουν το λόγο. Εάν όχι, ονόματο τη ομάδα μου των Πρασίνων. Θέλω να πω ότι ο Ρομπέρ μπορεί να είναι ικανός, πρέπει να είναι ικανοποιημένος γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο του James Bond και να πάει με αυτό στην Κορέα. Αλλά στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια μεγάλη ε, δυσκολία Ευρώπη με την εμπορική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ χρόνο δεν έχει υπογράψει εμπορική συμφωνία με την Κορέα και ένα <clears throat> από τα πρώτα παραδείγματα τέτοιων εμπορικών συμφωνιών θέτει ένα αμφιβόλο, ό,τι και να λέει η Κομισιόν, μία σαφή πολιτική για το περιβάλλον. Για μας αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό μήνυμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι φανερό ότι το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο θα εκπέμπεται από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα οποία χάρη στο λόμπι έχουν εξασφαλίσει μια αλλαγή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Κορέα, και εδώ και ένα θέμα αρχής. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση απέσπασε από την Κορέα την μείωση των φιλοδοξιών της για το περιβάλλον, τι θα γίνει με τις επερχόμενες συμφωνίες εμπορικού χαρακτήρα και φυσικά στα πλαίσια της αμεβαιότητας. Όταν έρθει ο Καναδάς και πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πούν ότι θέλουμε να αλλάξει μια ευρωπαϊκή οδηγία, χάρη για την ποιότητα των ε, καυσίμων, για να χρησιμοποιηθούν οι ασφαλτόδεις σχιστόληθοι του Καναδά, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πει όχι, γιατί είναι σημαντική η προτεραιότητα του περιβάλλοντος. Θα διατηρήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση την προσήλωση στο περιβάλλον και θα κρατήσει το περιεχόμενο της οδηγίας ή θα πει όπως είπε η Κορέα αφού αυτό αυξάνει τις εξαγωγές μας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας σε επίπεδο περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ νομίζουμε ότι έχει κάνει φάουλ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, που ενέπλεξε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια υποβάθμιση των προδιαγραφών του περιβάλλοντος στο βωμό τη πολιτική εμπορικών θεμάτων. Αυτό μα φαίνεται ότι είναι λάθο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώνει τι προσδοκίε τη για το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα και γι' αυτό εμεί σαν ομάδα θα καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία η οποία ανατρέπει μια ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέτει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρώτα και μετά μοναχά τα εμπορικά συμφέροντά της. Και δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει πει κάτι για να απαντήσει στους διάφορους παρεμβαίνοντες. Ναι, ναι. Να απαντήσω στα δύο ερωτήματα που έφυξε ο Παύλος Σάλβα και εσείς. Πρώτον, για το θέμα της, των προτύπων ασφαλείας. Όπως είπε και ο Παύλος Σάλβα, πραγματευθήκαμε με την Κορέα τέτοια πρότυπα από την αρχή. Και η Κορέα μας είπε ότι θέλει πλήρη ισοτιμία χωρίς κανένα περιορισμό των ευρωπαϊκών προτύπων. Αυτό καλύπτει όλα τα πρότυπα που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ως σημαντικά ως προς το κόστος της συμμόρφωσης και η Κορέα δέχεται ότι θα θεωρεί ασφαλές αυτό που θεωρείται ασφαλές και στην Ευρώπη χωρίς κανένα περιορισμό. Βεβαίως για άλλα πρότυπα θα χρειαστεί κάποια περίοδος πριν μπορέσει η Κορέα να εναρμονίσει την ομοθεσία της με την Ευρωπαϊκή. Αλλά όλα τα πρότυπα που μας ανέφερε η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία ότι δεν είναι προτεραιότητες θα μεταφερθούν εν καιρό το δέοντι. Επισήμως έχει υποσχεθεί η Κορέα ότι τα πρότυπα αυτά δεν θα αποτελέσουν η καθυστέρηση της εφαρμογής, δεν θα αποτελέσουν φραγμό για την πρόσβαση στην αγορά τους. Και γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι στη συμφωνία δεν υπάρχει τίποτα, ούτε στη συμφωνία της με τις ΗΠΑ που να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εις βάρος των Ευρωπαίων εξαγωγέων. Βέβαια επανέλαβα και ε, είπα και πριν ότι θα το προσέξουμε. Τώρα για το θέμα του κυρίου Γερό. Μπορώ να σας πω ότι η Κομισιόν συνεργά, εργάστηκε πολύ σκληρά συνεργασία με όλες τις αρμόδιες της υπηρεσίες και δεν ζήτησε ποτέ να μειωθεί το επίπεδο περιβαλλοντολογικής προστασίας της Κορέας. Δεν θέλουμε να μειωθούν τα πρότυπά τους και δεν επιβάλλουμε κανένα άδικο βάρος πρόσθετο στους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Είναι αναπόφευκτο η αρχική πρόταση των κορεατικών αρχών να έχει αλλάξει και να... Για οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο 6% της κορεατικής αγοράς. Απλώς θελήσαμε να μοιράσουμε αλλιώς το βάρος ώστε να μην το φέρουν όλο οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς. Ζητήσαμε εξισορρόπηση, νομίζουμε ότι επιτεύχθηκε και φυσικά αν θέλετε και άλλα σχόλια μπορώ να σας τα κάνω με τα χαράς, αλλά πάντως δεν έχει μειωθεί καθόλου η σημασία των υποσχέσεων που μας έδωσε η Κορέα. Η κατανομή του βάρους ήταν δίκαιη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο και σας υπενθυμίζω ότι πρέπει στις 5 να ψηφίσουμε, αλλά έχουμε ακόμα ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό για το Μαρόκο και υπάρχει και ένα σημείο ανταλλαγής απόψεων με την Κομισιόν, Γενική Διεύθυνση του Επιχειρήν, για το θέμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικών Οργανώσεων το να έχουμε ένα κέντρο πόρων και είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές εν ώψη τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που έχουμε για το θέμα αυτό και θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν να, να παρεύει ο Σεμπέρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κρίστιαν Ζίμπερτ λέγομαι, είμαι διευθυντής για τα γενικά θέματα στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Επιχειρήν. Οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πραγματικά πολύ δυναμικό για να διεισδύσουν σε τρίτες χώρες. Πολύ λίγες από αυτές το πράττουν όπως βλέπουμε και στις μελέτες μας. Χρειαζόμαστε πιο πολύ υποστήριξη και πληροφορίες και επίσης και μεγαλύτερες εταιρείε να μπορέσουν να ξενιτευτούν από ό,τι καταλαβαίνουμε και εργαζόμαστε με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις βιομηχάνων και επιχειρηματιών. Εδώ και πολύ καιρό έχουν κυρίως ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες αντιπροσωπείες μεγάλων επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν και εταιρείε που βρισκόνται σε τρίτες χώρες. Εμείς δεν τους χρηματοδοτούμε, αλλά ενθαρρύνουμε τη δραστηριότητά τους και τους προσκαλούμε δυο φορές το χρόνο σε συναντήσεις ώστε να αναπτύξουμε περισσότερο το δίκτυό τους και να έχουν επαφή με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν <clears throat> πολύτιμη εμπειρία αυτές οι οργανώσεις από τη δραστηριότητά τους σε τρίτες χώρες, από τις οποίες μπορεί να υποφελθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η εμπειρία βοηθά και τις ευρωπαϊκές εταιρείες, Ήδη στα θέματα της πρόσβασης σε αγορές τρίτων χωρών και των εμποδίων για αυτή την πρόσβαση. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ χρήσιμες για επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν την πρόσβαση σε τρίτες χώρες και τις υπηρεσίες της Κομισιόν που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Τώρα το δίκτυο των, ε, επιχειρήσεων θέλει να δημιουργήσει ένα γραφείο, να δημιουργήσει ένα γραφείο στην ε, Θεωρούμε ότι είναι συμπληρωματική αυτή η συλλογή πληροφοριών και παροχή πληροφοριών για τη γνώση των αγορών τρίτων χωρών, του επιχειρήν σε τρίτε χώρε κτλ. Όλα αυτά είναι συμπληρωματικά με αυτά που γνωρίζει η Κομισιόν. Η πρόσβαση στο δίκτυο λοιπόν επίση εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εκπροσώπων του είναι πολύ σημαντική και μα βοηθάει στη δημιουργία τη βάση δεδομένων για τα προσκόμματα σε <clears throat> δραστηριότητα σε τρίτε χώρε. Το δίκτυο αυτό λοιπόν να, η δημιουργία αυτού του δικτύου που περιλαμβάνει όλε αυτέ τι οργανώσει είναι ένα σημαντικό στόχο. Μερικέ από τι προτάσει που θα ανελάμβανε αυτό το, το δίκτυο θα μπορούσαν να επικαλύπτονται με δομέ ή με επιχειρήσει στα κράτη-μέλη και εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην χρηματοδοτήσουμε τέτοιε ενέργειε. Είναι ένα ανταγωνιστικό τομέα, και το να χρηματοδοτήσουμε ένα φορέα έχει επίπτωση και σε άλλου παίκτε στον τομέα αυτό. Επομένω πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Για το λόγο αυτό δεν έχουμε κάποια άποψη για την ετούμενη χρηματοδότηση, γιατί μια άμεση χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για άλλες επιχειρηματικές δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα τελευταίο στοιχείο σε σχέση με το γενικό πλαίσιο της εργασίας μας, η Κομισιόν προετοιμάζει μια ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο σε σχέση με την υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να θεσπίσει μια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτεραιότητες για την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τέτοιες πρωτοβουλίες. Η κοινοποίηση αυτή θα υπόκειται σε μια δημόσια διαβούλευση η οποία θα ξεκινήσει αν θέλει ο Θεός το Μάρτιο και μπορεί η ανακοίνωση αυτή να πάρει τελική μορφή το καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο. Η ανακοίνωση αυτή θα βασιστεί λοιπόν στα πορίσματα της μελέτης που έχει χρηματοδοτηθεί με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το δυναμικό της παγκοσμιοποίησης της δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για οι εμπειρίες που προέρχονται από τις πιλωτικές μελέτες έχουν και αυτές χρηματοδοτηθεί οι μελέτες με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα γραφεία υποστήριξης στην Κίνα και την Ινδία έχουν συμβάλει τα μάλα και η ανακοίνωση θα προτείνει κατευθυντήρε γραμμέ, όπω είναι παραδείγματο η ανάγκη συμπληρωματικότητα μεταξύ υπαρχουσών μορφών υποστήριξη και νέων μορφών υποστήριξη για τέτοιε υπηρεσίε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο, για τι πληροφορίε αυτέ και προφανώ θα λάβουμε υπόψη αυτέ τι πληροφορίε σε όλε τι συζητήσει που θα έχουμε για τα θέματα τη χρηματοδότηση και του προπολογισμού για να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να υποστηρίξουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε και πάλι μερσή. Οπότε προτού ξαναδώσω το, την προεδρία στον πρόεδρό μας, σας υπενθυμίσω ότι τώρα η συνεδρία είναι και κλεισμένων των θυρών. Μόνο σε αυτή την αίθουσα μπορούν να μείνουν οι κοινοβουλευτικοί, προφανώς, το προσωπικό της ε, Επιτροπής μας, οι συνεργάτες των πολιτικών ομάδων, οι προσωπικοί συνεργάτες των βουλευτών και η νομική υπηρεσία. Οι άλλοι λυπάμαι θα σας αποχωριστούμε.